Meine Κυρίες και κύριοι, κηρύσω την επανέναρξη της Συνόδου που διεκόπη στις 27 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως στις 27 Φεβρουαρίου είναι στη διαθέσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Κυρίες και κύριοι, η Ραζάμ Ζάιτσουνου ε, τιμηθήσαμε το βραβείο Ζαχάροφ πριν από δύο μήνες απήχθη μαζί με το σύζυγό της και ακόμη έναν ε, ε, αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα από μια ομάδα έξω από τη Δαμασκό δεν είναι γνωστό το που βρίσκεται. Τους τελευταίους δύο μήνες δεν έχουμε καμία είδηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τη ε, απευθύνει έκκληση για την ταχύτατη απελευθέρωση της κυρίας Τσουνή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε και αφιέρωσε τη ζωή του στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Έχει αντιμετωπίσει απειλές τόσο από το καθεστώς Συρίας όσο και από τις ομάδες των αντικαθεστωτικών αλλά δεν είναι και η μόνη η οποία έχει απαχθεί, βασανιστεί, κρατηθεί παράνομα. Είναι ένα ακόμα από τα θύματα των, του πολέμου αυτού. Πολλές φορές στη Συρία χρησιμοποιείται προκειμένου να καταπιεστεί περαιτέρω ο λαός, η κοινωνία της Συρίας ε, ως όπλο ο βιασμός. Πρέπει να τον καταδικάσουμε με κάθε τρόπο και πριν από δύο μέρες ξεκίνησε η σύνοδος για το θέμα αυτό. Πρέπει να τοποθετηθούμε, να υποστηρίξουμε άτομα και οργανώσεις που προστατεύουν και προσφέρουν βοήθεια στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού ώστε να μπορούν να ξαναγυρίσουν σε μια ομαλότητα στη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα και να καταγράψουν και να τεκμηριώσουν τα εγκλήματα αυτά που διαπράττονται. Άλλη μια φορά απευθύνουμε έκκληση για την απελευθέρωση της τιμηθής σας με το βραβείο Ζαχάροφ, και στις ανακοινώσεις. Η κυρία Φραντσέσκα Βαρατσού από τις 28 Φεβρουαρίου έχει αναλάβει καθήκοντα στην Ιταλική κυβέρνηση. κυβέρνηση. Ο κύριος Κλάους Χάινερ Λένε από 1η Μαρτίου 2014 ε, αναλαμβάνει καθήκοντα ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τους συγχαίρω και ενημερώνω σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού ότι σε σχέση με την κυρία Μπάρεμσο από τις 28 Φεβρουαρίου για τον κύριο Λένα από την 1η Μαρτίου χειρεύουν οι θέσεις τους. Δύναμη του άρθρου 74 του κανονισμού μας ε, έχω υπογράψει μία σειρά πράξεων μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και οι πράξεις αυτές θα προσερθούν στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης. Και προχωρώ στην ημερήσια διάταξη και τις αλλαγές της ή καλύτερα την έγκρισή της δυνάμει του άρθρου 137 ελήφθη απόφαση από το Προεδρείο, από τη των Προέδρων για την έγκριση για τον προσορισμό της ημερήσιας διάταξης στις 7 Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ορίζεται η ημερήσια διάταξη για την τρέχουσα σύνοδο και περνώ στην έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου, χαιρετίζοντα και τον κύριο Χόιε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η έκθεση, επενδύσεων, η έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου αφορά ακριβώς το θέμα της ετήσιας έκθεσης του 2012 για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ΕΤΕ γνώρισε μία αύξηση κεφαλαίου 10 δις ευρώ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μεταξύ 13-15 ε, θα φτάσει στα 60 δις για τη χρηματοδότηση μακροχρόνια.